Στρεβίτσιους. Κύριε Στρεβίτσιους, έχετε το λόγο. Mr. President. Κύριε Πρόεδρε, δυστυχώς έχει πολύ βαβούρα. So, Geschäftsordnung, Herr Kollege ναι, για διαδικαστικό θέμα κύριε Αυστρεβίτσιους, κύριε Πρόεδρε. Εάν βέβαια με ακούει κάποιος. Ακούστε παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, συνάδελφοι, πριν δύο χρόνια στις 2 Απριλίου 2014, εδώ, σε αυτό το σώμα, το Ευρωκοινοβούλιο, με απόλυτη πλειοψηφία υιοθετήσαμε μια σύσταση προς το Συμβούλιο για τη θέσπιση κοινών περιορισμών θεωρήσεων για Ρώσους αξιωματούχους που ήταν αναμειγμένοι στο θάνατο του Σεργέη Μαγνίτσκι. Σε αυτή τη σύσταση ε, ζητήσαμε από το Συμβούλιο, μεταξύ άλλων μέτρων, να εφαρμόσει και να ε, ε, ελέγξει την απαγόρευση ε, θεώρησης, έκδοσης θεώρησης σε 23 αξιωματούχους ε, υπεύθυνου για το θάνατο του Μαγνίσκη καθώς και υπεύθυνου για παρενόχληση της οικογένειάς του και της μητέρας του. Εχθές έγινε εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο μια εκδήλωση από έναν από τους συναδέλφους μας, ένα μέλος του Ευρωκοινοβουλίου από αξιοσέβαστη πολιτική ομάδα και επιστήνω την προσοχή στο γεγονός ότι λόγω αυτής της εκδήλωσης δύο άνθρωποι, δύο από τη λίστα Μαγνίσκη ήταν παρόντες ο Πάβελ Κάρποφ και ο Αντρέι Παύλοφ που ε, τους επιτρέπεται να έρθουν και να κάνουν και παρεμβάσεις. Ε, εκφράζω την λύπη μου ε, που έγινε κάτι τέτοιο εντός των τυχών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θέλω να επιστήσω την προσοχή σας στο πρόβλημα κύριε Πρόεδρε γιατί είναι θέμα ακεραιότητας των ίδιων μας των αποφάσεων. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ κύριε Αουστρεβούτσιος θα περάσουμε στη διαδικασία. Έχουμε μια πολύ μακρά διαδικασία ψηφοφοριών. Ε, οι υπηρεσίες μας έχουν, έχουν υπολογίσει ότι θα κρατήσει δύο ώρες και δεν θα γίνει λόγω αυτού του λόγου, λόγω αυτού του γεγονότος δεν θα γίνουν προφορικές επεξηγήσεις ψήφου παρά μόνο γραπτές. Ερχόμαστε λοιπόν στην ψηφοφορία. Η έκθεση ΆΣΙΣ, Συμφωνία για την Εναέριο Χώρο Ευρωπαϊκή Ένωση Γεωργία. Με ονομαστική κλίση άρχεται. Ψήφισατε όλοι. Ψήφισατε όλοι. Πέρας. Θέλει κάποιο το λόγο σε διαδικαστικό επίπεδο. Έχει γίνει δεκτή η, η συμφωνία αυτή. Κύριε Καβαντά, έχετε το λόγο. Δεν είναι διαδικαστικό, κύριε Πρόεδρε. Πρόκειται για ένα τεχνικό θέμα. Δεν ακούμε καλά την μετάφραση. Ο ήχος από την καμπίνα δεν είναι αρκετά δυνατός. Αν κάποιος τεχνικός μπορεί να το διορθώσει, θα ευχαριστήσουμε. Είναι ακόμα προβληματική η γαλλική μετάφραση. Εμένα μου φαίνεται κάπως καλύτερα να ακούγεται. Εντάξει. Περνάμε στη δεύτερη συμφωνία εκθεσιάσεις για την συμφωνία την Ευρωμεσογειακή με το Ισραήλ για τα αεροπορικά θέματα. Πάλι ονομαστική κλίση άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίθηκε. Έκθεση για κονσάρι. Συμφωνία για την αμοιβαία αρρωγή μεταξύ τελωνιακών αρχών. Έχει το λόγο η κυρία Γιακονσάρη για δύο λεπτά. Κυρία Γιάκονσάρη, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, Κοιτάξτε, τόσο θόρυβο ε, ε, επικρατεί εδώ μέσα που δεν άκουσα ότι μου δώσατε το λόγο. Θέλω να ευχαριστήσω του τελωνιακού υπαλλήλου εδώ Μιλάμε για την τελωνιακή συμφωνία ανάμεσα στην Κροατία και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι τελωνιακοί υπάλληλοι κάνουν πολύτιμο έργο για να εμποδίσουν την απάτη. Και θα πρέπει να εφαρμοστεί αυτή η συμφωνία όσο γίνεται πιο γρήγορα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κυρία Γιάκονσάρη. Ψηφίζουμε μονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Γίνεται δεκτή. Έκθεση Λεμπρετών για την ε, κοινοβουλευτική ασυλία του κυρίου Πίχα. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, έχει γίνει δεκτή. Ψήφισμα για την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού στην Ευρωπαϊκή Ένωση επί τη βάση των αιτήσεων που έχουν έρθει αναφρόπωθα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Υπάρχει τώρα αιτήση διαβούλευση Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής υπέρ, κατά, αποχές, Εγκρίθηκε. Έρχομαι στην έκθεση Τσίλε για την ε, Σιδηροδομική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κοινή θέση, πρόταση απόρριψης θέσης του Συμβουλίου υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Επομένως έχει γίνει δεκτή η κοινή θέση και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έκθεση Μπιλμπάο παρα, παραντικά πάλι πρόταση για την απόρριψη της θέσης του Συμβουλίου ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται και αυτή και πάλι η νομική αυτή πράξη με τη Συμφωνία Συμβουλίου και Κοινοβουλίου έχει γίνει δεκτή. Έκθεση Κράμερ. Πάλι πρόταση για την απόρριψη της θέσης του Συμβουλίου ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Επομένως και σε αυτήν την περίπτωση διαπιστώνω ότι η συμφωνία του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ισχύει. Θέλετε επαλήθευση βεβαίως. Άρχεται η επαλήθευση ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Έχει γίνει λοιπόν η ισχύ συμφωνία Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Αρχόμαστε στην έκθεση Νιούβενχέιζεν. Το σύνορο ο, και εδώ η εισηγητής έχει το λόγο για δύο λεπτά. Η κυρία εισηγητή έχει το λόγο για δύο λεπτά. Μικρόφωνο, πείτε. Μικρόφωνο, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι μπορούμε να είμαστε όλοι περήφανοι για την Ευρώπη που θα είμαστε οι πρώτοι στον κόσμο που έχουμε νομοθεσία για να αποφεύγουμε χειραγώγηση σημαντικών δικτών όπως το Λάιμπορο κλπ. Αυτό γίνεται εξαιτία τη καλή δουλειά που κάναμε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θέλω να ευχαριστήσω τον Τούλμαν Ντεμαέρα, τον Φερνάντε, Κέι Σουίπερτ και όλο το προσωπικό που βοήθησε στην εκτέλεση αυτού του έργου. Σα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Φανίου Ενχόιζεν. Τροπολογία 2. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Πρόταση της Κομισιόν. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές γίνεται δεκτή. Ψη, νομοθετικό ψήφισμα με ονομαστική κλίση άρχεται η, ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται. Έκθεση τη Λαπάγιοβα για την απαλλαγή 2014 ε, το, η απόφαση σας σύνολο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Στο ψήφισμα τώρα. 21 υπέρ κατά αποχές την Τροπολογία 49 υπέρ. Κα... Θέλετε έλεγχο στην 21. Μάλιστα, άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Απορρίφθηκε 21. 49 υπέρ. Κατά αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά σε ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Παράγραφος 66, το αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά αποχές δεκτό. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά. Θα ελέγξουμε για το δεύτερο τμήμα άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Παράγραφο 68 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 24 υπέρ. Έλεγχος για την 23. Άρχεται η ψηφοφορία. Ελέγχουμε για την 23. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. 24 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 25 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 26 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 4 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 5 με ονομαστική κλίση. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 50. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 27. 50 έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Haben alle abgestimmt? Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτηκε. 27. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 51. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 52. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 6 υπέρ <clears throat> κατά αποχές απορρίπτεται 8 με ονομαστική κλίση άρχεται Σφίσατε όλοι πέρας απορρίπτεται 9 με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία Σφίσατε όλοι πέρας Εγκρίνεται. 10. Με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίθηκε. 28. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 58. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 29 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Παράγραφος 243 το αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 53. Ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. 54 πάλι μονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισατε όλοι. Πέρας. μου. Τροπολογία 3 σε δύο τμήματα. Η τροπολογία 3 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα ονομαστική κλίση άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Δεκτό. Δεύτερο τμήμα, πάλι μονομαστική κλίση, άρχεται. Ψήφισατε όλοι. Πέρασε. Εγκρίθηκε. 55 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 30 με 35 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 36 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 37 υπέρ 36 έλεγχος άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία ψηφίσατε όλοι πέρας εγκρίνεται 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 39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 αποχές απορρίπτεται. 43 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 44 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 45 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 46 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 11 με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. 46 έλεγχος προηγουμένως, ηλεκτρονικά, άρχεται. Ψηφίσατε όλοι, πέρας. Απορρίπτεται με ψηφία. 11 με ονομαστική κλίση. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απολύτωται. 47 μονομαστική κλίση άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. 57 ονομαστική κλίση άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Εκπίπτει το αρχικό κείμενο. Τροπολογία 12 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 48 σε τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. Δεύτερο τμήμα έλεγχος. Άρχεται. Φυσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Τρίτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Αρχικό κείμενο της 400. Ψήφι υπέρ. Κατά. Δεν είναι σαφές. Φαντάζομαι ότι απορρίπτεται, αλλά κάνουμε έλεγχο. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 405 το αρχικό κείμενο μονομαστική κλίση αρχίζει. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας Ψηφοφορίες. Εγκρίνεται. Παράφος 410 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 434 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογίες 13 και 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. Συγγνώμη, συγγνώμη. Φυσικά απορρίπτονται. 15. Υπέρ. Έκανα λάθος. Ήταν γλωσσικό. 15. Ε, υπέρ. Κατά. Αποχές. απορρίπτεται. 16. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 17. Υπέρ κατά αποχές 18 σε δύο τμήματα ονομαστική κλίση πρώτο τμήμα άρχεται ψήσατε όλοι πέρας απορρίπτεται δεύτερο τμήμα με ονομαστική κλίση πάντα άρχεται ψήφισατε όλοι πέρας και αυτό απορρίπτεται. 19 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 20 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Το σύνολο με ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. πέρας. Εγκρίνεται. Και μία ακόμα έκθεση Λαμπαγιώβα, η ειδική έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου, το αρχικό κείμενο, παράγραφος 9, μονομαστική κλίση, άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Συγγνώμη. Άρχεται η ψηφοφορία και πάλι. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Το σύνολο του ψηφίσματος με ονομαστική κλίση και πάλι άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Ερχόμαστε. Στην έκθεση Σμιτ απαλλαγή για το 8ο, 9ο, 10ο και 11ο πρόγραμμα ε, αναπτυξιακού χαρακτήρα. Άρχεται η απόφαση με ονομαστική κλίση. Ψηφίζουμε. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται για το ψήφισμα. Τροπολογία 2 υπέρ. Κατά Αποχέ. εγκρίνεται. 8 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 79 το αρχικό κείμενο. Υπέρ. Κατά απόχέ εγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ. Κατά Αποχέ εγκρίνεται. Τροπολογία 1 με ονομαστική κλίση. Έλεγχος για την τρία, μάλιστα. Ξεκινάμε. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτωτε. Τροπολογία 1 με ονομαστική κλίση άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τέσσερα μονομαστική κλίση. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Πέντε μονομαστική κλίση. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Παράγραφος 100 το αρχικό κείμενο. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Έξι μονομαστική κλίση άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. 7. Ονομαστική κλίση. Άρχεται. Ψήφισατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Ε, εκπίπτει το αρχικό κείμενο και πάμε στο σύνολο λοιπόν με ονομαστική ψηφοφορία. Το σύνολο του κειμένου. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Έκθεση Πίπερ. Απαλλαγή 2014 για το Γενικό Προπολογισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Παρακαλώ για διαδικαστικό έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Παράγραφος 49 που αφορά την απαγόρευση παρά, παρά, ε, δεύτερες δουλειές για τους ευρωβουλευτές. Εγώ θέλω να... Μάλλον ζητήθηκε χωριστή ψηφοφορία πολύ μετά την ημερομηνία προθεσμίας. Πιστεύουμε πως είναι απαράδεκτο αυτό το αίτημα για ε, κατατμήματα ψηφοφορία που ζητήθηκε μετά από την λήξη της προθεσμίας για τόσο σημαντικό θέμα παρότι ο πρόεδρος Σουλς το ενέκρινε. Ζητώ λοιπόν να μην ψηφιστεί. Αν όμως ε, θεωρείται εξαιρετική διαδικασία και γίνει τέτοιου είδους ψηφοφορία, θέλουμε να γίνει ε, ονομαστική κλίση. Ευχαριστώ. Mir wird gesagt, dass der Präsident das entschieden hat, dass man darüber abstimmt. Εάν ο πρόεδρος έχει, αποφάσεις, έχει αποφασίσει να ψηφιστεί αυτή η παράγραφος. εγώ δεν μπορώ να αλλάξω αυτή την άποψη καταγράφω ότι ζητήσατε ονομαστική κλίση απλώ και μόνο. Θα το κάνουμε αυτό. Ξεκινάμε με την απόφαση για το σύνολο της απαλλαγής. Ναι. Υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. Για την, το ψήφισμα. Παράγραφος 13. Το αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχέ δεκτό. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχέ απορρίπτεται. Παράγραφος 14. Αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται δεύτερο τμήμα υπέρ Εκπίτω το δεύτερο τμήμα παράγραφος 18 τροπολογία 14 ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται παράγραφος 23 αρχικό κείμενο με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία ψηφίσατε όλοι πέρας εγκρίνεται Παράγραφος 26 αρχικό τμήμα σε δύο, σε τμήμα. Πρώτο τμήμα. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν βλέπω κανένα να ψηφίζει από τα δεξιά μου. ότι ε, κάνουμε επαλήθευση για το δεύτερο τμήμα. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 5. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 32 το αρχικό κείμενο υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 37 έχει αποσυρθεί. 58 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. εγκρίνεται. Οπότε εκπίπτει η 57 και το αρχικό κείμενο. 34 μονομαστική κλίση άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. 59 μονομαστική κλίση άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας εγκρίνεται, οπότε εκπίπτει και η 40. Παράγραφος 36, το αρχικό κείμενο μονομαστική κλίση άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 37, αρχικό κείμενο μονομαστική κλίση άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. 60 με ονομαστική κλίση. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Εκπίπτουν οι 44 και 45. Πάμε στη 15. Υπέρ. Κατά. Γιατί δεν, ε, δεν ψηφίζουν οι σοσιαλιστές κατά. Αποχές απορρίπτεται. 31 με ονομαστική κλίση. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. 32 με ονομαστική κλίση. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 7 με ονομαστική κλίση ξεκινά ψηφίσατε όλοι τελείωσε η ψηφοφορία εγκρίθηκε τροπολογία 1 πάλι με ονομαστική κλίση ξεκινάμε ψηφίσατε όλοι τέλος Εγκρίθηκε. 33. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 16 και 34 που είναι ταυτόσιμες σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα ονομαστική κλίση ξεκινάει η ψηφοφορία. Ψήφισατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος της προφορίας. Απορρίπτεται. 35 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Εκπίπτει 17 επομένως. Παράγωφο 49 αρχικό κείμενο. Ζητήθηκε ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισατε όλοι. Τέλος της προφορίας. Απορρίπτεται. 53 το αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 46 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 47 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Έλεγχος για τη 47. Ξεκινάει η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Δύο με ονομαστική κλίση άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Τρία μονομαστική ψηφοφορία. Ξεκινά. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 8. Άρχεται η ψηφοφορία. Συγγνώμη. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 20 και 21. Καθώς και 48 που είναι ταυτόσιμες. Με ονομαστική κλίση Ξεκινάει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτονται. 36 με, με προφορική τροπολογία από τον κύριο Πίπα. Κύριε Πίπα. Μικρόφωνο παρακαλώ κύριε Πίπερ. Πρόκειται για την τροπολογία για το βραβείο Λουξ. Θέλουμε να διαγράψουμε. Πρόκειται για μια μελέτη η οποία δεν είναι διαθέσιμη αυτή τη στιγμή. Λέει το κείμενο. Λυπάται πάρα πολύ ότι η μελέτη αυτή δεν είναι διαθέσιμη. Θέλουμε να διαγράψουμε το δίπλη ότι λυπούμαστε βαθιά ότι δεν είναι διαθέσιμη και επίσης πρέπει η έκθεση αυτή να δοθεί στην Επιτροπή Κουλτ, Επιτροπή Πολιτισμού και όχι μονάχα στην Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού. Αυτή είναι η προφορική τροπολογία τεσσάρων πολιτικών ομάδων. Υπάρχουν αντιρρήσει. Όχι. Τι ψηφίζουμε λοιπόν με αυτή τη διατύπωση υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 22 και 49 που είναι ταυτόσιμε, ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα τη πληροφορία. Εγκρίνεται. 72 αρχικό κείμενο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 73 αρχικό κείμενο με ονομαστική κλίση ξεκινάει η ψηφοφορία. Όλοι ψηφίσατε. Πέρας. Εγκρίνεται. 50 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 75. Αρχικό κείμενο με ονομαστική κλίση άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. 25 με ονομαστική κλίση. Ξεκινούμε. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος της απορρίπτεται 51 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται έλεγχος για την 51 ξεκινάει η ψηφοφορία επαλήθευσης Σφίσατε όλοι πέρας απορρίπτεται 83 το αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. 84 αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά αποχέ εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά απόχέ εγκρίνεται. 85 αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά αποχέ εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχέ απορρίπτεται. Τροπολογία 29 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 9 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 18 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 26 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται πράφος 99 αρχικό κείμενο με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία ψηφίσατε όλοι πέρας απορρίπτεται 52 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά <clears throat> αποχές απορρίπτεται 27 με ονομαστική κλίση ξεκινούμε ψηφίσατε όλοι τέλος της προφορίας απορρίπτεται 4 με ονομαστική κλίση αρχίζει η ψηφοφορία ψηφίσατε όλοι Τέλος προφορίας. Απορρίπτεται. 13. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 61 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 28. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται αρχικό κείμενο 126 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ σοσιαλιστές που είναι υπέρ πάλι <clears throat> κατά αποχές θα το ελέγξουμε το ελέγξουμε σας παρακαλώ με τον τρόπο αυτό καθυστερούμε άμα δεν σηκώνετε τα χέρια σας μια ολόκληρη ομάδα δεν ψηφίζει λοιπόν ψηφίσατε όλοι πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 54 <clears throat> υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 55 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 56 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 19 υπέρ κατά ελέγχουμε την 19. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψήφισατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. 135 το αρχικό κείμενο σε με τα πρώτα τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 11 ονομαστική κλίση ξεκινάμε. Όλοι ψηφίσατε πέρας απορρίπτεται 12 ονομαστική κλίση ξεκινάμε ψηφίσατε όλοι πέρας απορρίπτεται το σύνολο του ψηφίσματος με ονομαστική κλίση άρχεται η ονομαστική κλίση ψηφίσατε όλοι πέρας Εγκρίνεται. Έκθεση Τσανέσκη. Προπολογισμό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο. Απόφαση για την αναβολή τη ε, ε απαλλαγή σε ονομαστική κλίση. Άρχεται. Ψήφισατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Το ψήφισμα σύνολο πάλι με ονομαστική κλίση άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Έκθεση φίστησεν. Η απόφαση σαν σύνολο ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Το ψήφισμα. Τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. απόχέ Απορρίπτεται. Τροπολογία 2 υπέρ. Κατά. απόχέ Απορρίπτεται το σύνολο με ονομαστική κλίση άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Έκθεση Τσανέσκη για το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Απόφαση για την απαλλαγή ψήφι υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Ψήφισμα τροπολογία 1 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Το σύνολο του ψηφίσματος με ονομαστική κλίση άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Έκθεση βίστησεν για την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Η απόφαση καταρχήν ο σύνολο ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Το ψήφισμα τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά αποχές ελέγχουμε για, το, για την τροπολογία 1. Άρχεται η ψηφοφορία. Με μεγάλα κομμάτια της Ολομέλης δεν ψηφίζουν δυστυχώς. Πέρασε ψηφοφορίες. Εγκρίνεται. Δεύτερη. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχέ απορρίπτεται. 4. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Έλεγχο για το 4. Άρχεται η ψηφοφορία έλεγχου. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας τη προφορία. Εγκρίνεται. Το σύνολο του ψηφίσματος με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ονομαστική κλίση. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα. Εγκρίνεται. Έκθεση Μακοβέη για την Επιτροπή των Περιφερειών η απόφαση απαλλαγή ψήφι υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. Το ψήφισμα τώρα τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται έλεγχος για το 1 <clears throat> άρχεται η ψηφοφορία ψηφίσατε όλοι πέρας απορρίπτεται τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 3 υπέρ κατά Ελέγχουμε την 3. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Έγκρινεται. 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 5. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Κάνουμε έλεγχο και για την 5. Άρχεται η ψηφοφορία ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Η 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Εκπίπτει η 7 ως εκ τούτου. Το σύνολο του ψηφίσματος ρωμαστική κλίση ξεκινάμε. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκέκριται. Έκθεση αρνεύσης για την ε,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 Τροπολογία 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Παράγραφος 27 αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά <clears throat> αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 5 υπέρ. Θέλετε έλεγχο για την ένα, βεβαίως. Άρχεται η ψηφοφορία έλεγχο. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 5 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Έξι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Το σύνολο του ψηφίσματος μονομαστική κλίση άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίθηκε. Έκθεση Τσαρνέσκη για την διαμεσολαβήτρια. Η απόφαση ο σύνολο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το ψήφισμα τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές κάνουμε έλεγχο στην 2 ε, άρχεται η ψηφοφορία Φύσατε όλοι πέρας ψηφοφορίας Γκρίνεται Τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος για την 3. Άρχεται η ψηφοφορία έλεγχος. όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. 4 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 5. Με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Παράγραφος 22. Το αρχικό κείμενο με ονομαστική κλίση. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται το σύνολο του ψηφίσματος. Μονομαστική κλίση ξεκινάμε. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίθηκε. Έκθεση Μακοβέη για τον Ευρωπαϊκό Επόπτη για τα ε, προσωπικά στοιχεία. Η απόφαση έχει γίνει δεκτή. Το ψήνο... Άρχεται η ψηφοφορία για το ψήφισμα. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Πολλές εκθέσεις, εκθέσεις του κυρίου Βόν τώρα. Η πρώτη είναι για την απόδοση, την οικονομικό έλεγχο των ε, αποκεντρωμένων φορέων. Παράγραφος 18, τροπολογία 2, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 1, υπέρ, 2, ελ, υπέρ. Συγγνώμη. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά για τη δύο Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Το ψήφισμα σύνολο. Ονομαστική ψηφοφορία άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Η Υπηρεσία για τη Συνεργασία των Ρυθμιστών Ενέργειας. Απόφαση για την απαλλαγή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ψήφισμα ως σύνολο με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίθηκε. Πάλι εκτεσιβών το γραφείο των ρυθμιστών για τα ηλεκτρικά θέματα η απόφαση ως σύνολο ψηφιπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το ψήφισμα με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. <clears throat> Εγκρίνεται πάλι βόν το κέντρο μετάφραση των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η απόφαση ως σύνολο ψηφιπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το ψήφισμα σε ονομαστική κλίση άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίθηκε. Έκθεση Βον Σέντεφοπ, Κέντρο για την Ανάπτυξη Επαγγελματική. Η απόφαση υπέρ κατά δεκτή το ψήφισμα σύνολο με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίθηκε. Βον για το ΣΕΠΟΛ η απόφαση στο σύνολο ψήφι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Το ψήφισμα με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Η Υπηρεσία Αεροπορικής Ασφάλειας, ΕΑΣΑ, η απόφαση στο σύνολο υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Το ψήφισμα με ονομαστική κλίση άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Βόν Υπηρεσία ε, Υποστήριξης Ασύλου ΕΑΣΟ, η απόφαση ο σύνολο υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, το ψήφισμα με ονομαστική κλίση άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή. Η απόφαση απαλλαγής υπέρ, κατά, αποχές δεκτή το ψήφισμα μονομαστική ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Βον. εδώ για την πρόληψη των ασθενειών. Η απόφαση ως σύνολο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το ψήφισμα μονομαστική ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισατε όλοι. Πέρας. Εγκρίθηκε. Βον Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για τα Χημικά η απόφαση απαλλαγής υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε το ψήφισμα με κλίση άρχεται. <clears throat> Ψήφισατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Βον Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος απόφαση υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε το ψήφισμα με ονομαστική κλίση άρχεται. Ψήφισατε όλοι. Πέρας. Εγκρίθηκε. Υπηρεσία για τον έλεγχο των αλλιευμάτων. Απόφαση απαλλαγής υπέρ κατά αποχές δεκτή. Παράγραφος 23 το αρχικό κείμενο υπέρ κατά αποχές εγκρίθεται τελικό ψήφισμα υπέρ μονομαστική κλίση άρχεται ψηφοφορία. Ψήφισατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Βον. Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Τροφιμικής Ασφάλειας. Η απόφαση ως σύνολο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το ψήφισμα. Τροπολογία 3. Έλεγχος για την απόφαση ως σύνολο. Άρχεται η ψηφοφορία. Πάει ίσως πιο γρήγορα έτσι. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Παράγραφος 8 αρχικό κείμενο σε τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Συγγνώμη. Εγκρίνεται το πρώτο τμήμα, λέει ο Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τρίτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Μάλλον απορρίπτεται. Κάνουμε έλεγχο για το 3. Ηλεκτρονικά άρχεται. Ψήφισατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Τρο, τροπολογία 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 5 με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. 6. Μονομαστική κλίση. Άρχεται. Ψήφισατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Παράφος 11. Το αρχικό κείμενο υπέρ. Κατά. Αποχέ. εγκρίνεται. Τροπολογία 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 13. Αρχικό κείμενο υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 8 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται, τροπολογία 1 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται, τροπολογία 2 υπέρ, <clears throat> κατά, αποχές απορρίπτεται, το σύνολο του ψηφίσματος, ονομαστική κλίση, ξεκινάμε. Ψηφίσαμε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Έκθεση Βον, Ινστιτούτο Ισότητας των Φύλων. Απόφαση, ψήφι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Ψήφισμα, ονομαστική κλίση άρχεται. Ψηφίσαμε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. <clears throat> Έκθεση Βον, ΕΙΟΠΑ. Συντάξεις και τέτοια θέματα. Απόφαση, ο σύνολο υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Ψήφισμα, ονομαστική κλίση. Ξεκινάμε. Ψήφισαμε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Βον. Ίδρυμα Τεχνολογίας και Καινοτομίας στο σύνολο της απόφασης υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ψήφισμα ο σύνολο με ονομαστική κλίση άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Οργανισμός φαρμάκων υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Ονομαστική ψηφοφορία, το επόμενο, α, μια στιγμή. Παράγραφος 20 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Τώρα το σύνολο του ψηφίσματος, ονομαστική ψηφοφορία, ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι, πέρασε τη ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Βόαν πάντα παρατηρητήριο τοξικομανίας. Η απόφαση υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ψήφισμα με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Βον πάντα. Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Αναφυλακής Ασφάλειας. Απόφαση υπέρ, κατά, αποχές, Εγκρίνεται. Ψήφισμα με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέραστη της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Βον, πάντα Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών. Απόφαση υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Ψήφισμα με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας της φοφορία. Εγκρίθηκε. Βον, πάντα Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ιδηροδρόμων. Απόφαση υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Ψήφισμα με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Βον, έσμα, απόφαση υπέρ, κατά, αποχές Εγκρίνεται. Ψήφισμα με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίστε. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματική Εκπαίδευση. Απόφαση υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. Ψήφισμα με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα τη ψηφοφορία. Εγκρίθηκε. Βόχαν πάντα, Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Διελεκτρική Διαχείριση, Λίζα. Απόφαση υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, ψήφισμα με ονομαστική ψηφοφορία, ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα τη ψηφοφορίες. Εγκρίνεται. Τώρα, ευρωπαϊκός οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία. Απόφαση υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Ψήφισμα με ονομαστική ψηφοφορία. Μπορείτε να ψηφίσετε. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε τη ψηφοφορία. Εγκρίθηκε. Οργανισμός ε, τη ΕΖΑ υπέρ εγκρίνεται. Ονομαστική ψηφοφορία για το ψήφισμα. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε τη ψηφοφορία. Εγκρίθηκε. Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθήκων Διαβίωση Εργασία. Απόφαση υπέρ, κατά, αποχέ εγκρίνεται. Ψήφισμα με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα τη ψηφοφορία εγκρίνεται. Μονάδα δικαστική συνεργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Eurojust, απόφαση υπέρ, κατά απόχέ εγκρίνεται. Ψήφισμα με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίθηκε. Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία Europol. Απόφαση υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Το ψήφισμα με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίθηκε. Οργανισμός Θεμολογιών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απόφαση υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ψήφισμα. Α, δύο Υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. Το ένα καταπίπτει. Πρόταση ψηφίσματος. Τώρα με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Frontex. Τώρα η απόφαση υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και το ψήφισμα, ονομαστική ψηφοφορία, ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίθηκε. Τέλος, για τον ΠΟΧΑΝ, Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή του Παγκόσμιου Δορυφορικού Συστήματος Πλοήγησης, απόφαση υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το ψήφισμα τώρα, ονομαστική ψηφοφορία, ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα στις φοφορίες. Εγκρίνεται. Τώρα, περνάμε. Δεν τελειώσαμε. Περιμένετε, περιμένετε. Μαρινέσκου τώρα αρχίζουμε. Ενσωματωμένα συστήματα υπολογιστών πρώτα, Άρτεμις. η απόφαση υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ψήφισμα, ονομαστική ψηφοφορία ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα τη ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Τώρα, κοινή επιχείρηση Clean Sky. Απόφαση υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ψήφισμα, ονομαστικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα τη ψηφοφορία εγκρίθηκε. Κοινή επιχείρηση ECSEL. Απόφαση υπέρ. Όχι, ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ, ηλεκτρονικά ψηφίζουμε. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα τη ψηφοφορίες. Εγκρίθηκε. Τώρα το ψήφισμα, πάλι με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι, πέρα τη ψηφοφορία. Εγκρίθηκε. Κοινή επιχείρηση ΕΝΙΑΚ. Απόφαση. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ψήφισμα στο σύνολό του τώρα, υπέρ. Να μάλλον ονομαστικά ψηφίσατε όλοι. Πέρα τη ψηφοφορία. Εγκρίθηκε. Κοινή επιχείρηση Κυψέλης Καυσίμου και Υδρογόνου. Απόφαση υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ψήφισμα ονομαστικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα της πουφορίας. Εγκρίθηκε. Κοινή επιχείρηση πρωτοβουλία για καινοτόμα φάρμακα 2. Απόφαση υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το ψήφισμα τώρα ονομαστικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα της φοφορίας. Εγκρίθηκε. Κοινή επιχείρηση για τον ΙΤΕΡ, για ανάπτυξη πυρηνικής σύνδεξης. Απόφαση για αναβολή της απαλλαγής. Ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα της φοφορίας. Εγκρίθηκε. Τώρα, πρόταση ψηφίσματο. Παράγραφος 3. Αρχικό κείμενο, δύο τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, απόχέ, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 1. Με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας τη ψηφοφορία. Απορρίφθηκε. Παράγραφος 5. Αρχικό κείμενο. Τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. απόχέ. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα υπέρ. Κατά. αποχέ. Εγκρίνεται και τώρα το ψήφισμα στο σύνολό του, τροποποιημένο βέβαια, με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι πέρα τη ψηφοφορία εγκρίθηκε. Κοινή επιχείρηση Σέζαρ. Πρόταση υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ψήφισμα, ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Ερχόμαστε τώρα στην έκθεση Πυρίνσκι. Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Ετήσια έκθεση 2014. Τροπολογία 7. Ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Παράγραφος 9. Αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 39. Παράγραφος 2 τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Παράγραφο 40, δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, νομίζω εγκρίνεται. Να ελέγξουμε. Ωραία, θεύουμε για το πρώτο τμήμα της παραγράφου 40. Ψηφίστε. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα της φοφορίας. Απορρίφθηκε. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Α, και εδώ θέλετε να επαληθεύσουμε. Ωραία. Ψηφίστε παρακαλώ ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα στις ψηφοφορίες. Εγκρίθηκε. Τρίτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. Παράγραφος 54, δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχέ εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχέ εγκρίνεται. Παράγραφος 59, αρχικό κείμενο υπέρ, κατά, αποχέ εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο 41, τροπολογία 1 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 2 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 3 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 5 υπέρ, σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές θα παληθεύσουμε. Πρώτο τμήμα της τροπολογίας 5. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα της ψηφοφορίας. εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται με την ίδια πλειοψηφία, πιστεύω. Αν θέλετε, επαληθεύουμε. Ωραία, ηλεκτρονικά ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας της προφορίας. Εγκρίθηκε. Έξι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη ε, αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα, καταπίπτει. Το σύνολο του ψηφίσματος τώρα με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στις προτάσεις ψηφίσματος σχετικά με τις επιθέσεις σε νοσοκομεία και σχολείο ως παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Έχουμε πρόταση ψηφίσματος κοινή 7 πολιτικών ομάδων υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται 5 σε δύο τμήματα με ονομαστική ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα υπέρ, μάλλον ονομαστικά ψηφίσατε όλοι πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Δεύτερο τμήμα. Ψηφίστε ονομαστικά πάντα. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα τη φοφορία. Εγκρίθηκε. Τρίτο τμήμα. Ψηφίστε παρακαλώ, ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα τη φοφορία. Εγκρίθηκε. Τέταρτο τμήμα. Ψηφίστε. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. 10. Παράγραφο σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχέ, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά, αποχέ, εγκρίνεται. 11. Αρχικό κείμενο σε ονομαστική κλίση, άρχιδη ψηφοφορία. Ψ, ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. 6 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Απορρίπτεται, συγγνώμη. 21 αρχικό κείμενο με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. Αιτιολογική σκέψη G σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 3 με ονομαστική κλίση άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Το σύνολο του ψηφίσματος υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Εκπίπτουν τα άλλα ψηφίσματα. Έκθεση Φεράρα πρόσβαση στα δημόσια έγγραφα για το 2014-2015. Τροπολογία 7, Πρώτο, δύο τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά, εγκρίνεται. Παράγραφος 8 σε δύο τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Ναι, δεν ναι, θέλετε έλεγχο, σωστό. Πρώτο τμήμα άρχεται η ψηφοφορία ελέγχου. Ψήσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίθηκε. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίθηκε. 9 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίθηκε. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίθηκε. Πράφος 10 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 14 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Παράφος 15 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 24 υπέρ. Έλεγχος για το δεύτερο τμήμα της 15 μάλιστα. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 24 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 25 σε δύο κομμάτια. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 27 σε ονομαστική ψηφοφορία. Τροπολογία 1, μάλιστα, ονομαστική ψηφοφορία άρχεται. Ψηφίσατε όλοι, πέρας. Αποδίδεται. Παράγραφος 29. Αρχικό τμήμα σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. 31. Δεύτερο τμήμα έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεν είναι εύκολο να βλέπω. Μερικές φορές δεν σας βλέπω. Τροπολογία 31. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Και τώρα το ECR δεν ψηφίζει. Πάλι 31. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 33 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο, μονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. 34 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 40. Πάλι σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 42. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Το σύνολο του ψηφίσματος. <clears throat> Θέλετε έλεγχο 42-2. Άρχεται η ψηφοφορία. Mm. Πέρας θα ήθελα να πω ότι όλες οι ομάδες πρέπει να ψηφίσουν, εγκρίνεται το σύνολο του ψηφίσματος, μονομαστική κλίση άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται. Έκθεση Κούνεβα για τις γυναίκες τις οικιακές υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση πως ένα Ονομαστική κλίση άρχεται. Ψηφίστε. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράφος 2 στα 4. Αρχικό κείμενο. Πρώτο τμήμα. Πάντα με ονομαστική κλίση. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, <clears throat> μάλλον άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Τρίτο τμήμα. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. εγκριτ Τέταρτο τμήμα. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας εγκρίνεται. Παράγραφος 9 αρχικό κείμενο υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 11 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Παράγραφος 12 με ονομαστική κλίση άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 13, ονομαστική κλίση άρχεται. Ψήσατε όλοι. <clears throat> Πέρας. Εγκρίνεται. 14 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 17 στα 3. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 19 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Παράγραφος 22 σε τρία τμήματα με ονομαστική κλίση κάθε φορά. Πρώτο τμήμα άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Τρίτο τμήμα. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 23. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. 24. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 25. Με ονομαστική κλίση. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται. 32. Υπέρ κατά Αποχέ, εγκρίνεται 33 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ Αποχέ, δεκτό δεύτερο τμήμα ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία ψηφίσατε όλοι πέρας εγκρίνεται 34 υπέρ κατά παρακαλώ 34 ψηφίστε υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται 35 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 41 υπέρ 40 μάλλον υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 41 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 43 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 56 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ <clears throat> κατά αποχές απορρίπτεται. 60 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 61 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 64 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά πολλές αποχές. Θα ελέγξουμε πρώτο τμήμα του 64. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Η διαπλειοψηφία εγκρίνεται. 65. Υπέρ. Κατά η ίδια πλειοψηφία νομίζω εγκρίνεται 66 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 68 υπέρ έλεγχος για την 66 άρχεται η ψηφοφορία ψηφίσατε όλοι πέρας απορρίπτεται Υπήρξαν πολλές, ε, πολλοί που δεν ψήφισαν, 68 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη έψεω σε τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τρίτο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Αιτιολογική σκέψη Α, λατινικό. Έλεγχος για το τρίτο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη I. Σε τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τρίτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη K. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Αιτιολογική σκέψη Ο. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Δεύτερο υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Αιτιολογική σκέψη R. Υπέρ. Έλεγχος στο δεύτερο τμήμα της αιτιολογικής σκέψης Ο. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφιστε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Αιτιολογική σκέψη R. Υπέρ. Κατά. Δύο ομάδες δεν ψηφίζουν. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε ψηφοφορίες, λέει ο πρόεδρος. Έγκριεται. Αιτιολογική σκέψη V, Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Y. Αιτιολογική σκέψη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη Z σε δύο. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Απορρίπτεται μάλλον. Αιτιολογική σκέψη ΑΕ. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. AG υπέρ Έλεγχος δεύτερο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. AG υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. AH υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. AI υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. AK υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. AM σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά δεκτό. Δεύτερο τμήμα υπέρ <clears throat> κατά αποχές απορρίπτεται. AO συγγνώμη. AM δεύτερο τμήμα έλεγχος αρχής ψηφοφορία ελέγχου. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απολύτωται. AO σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. AX <clears throat> υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. BA υπέρ. Κατά. Αποχές. Απολύτωται. BD σε ονομαστική κλίση. Άρχεται ψηφοφορία. Ψήφισατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη B υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. BF υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. BL σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. BM υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται το σύνολο με ονομαστική κλίση άρχεται. Ψήφισατε όλοι. Πέρας. Εγκρίθηκε. Τελευταία και τυχερή έκθεση, η έκθεση Ράιντχε ισότητα ανδρών και γυναικών στην ψηφιακή εποχή. Παράγραφος 9 αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 10 αρχικό κείμενο. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Παράγος 11. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. Παράγος 15. Δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. Παράγος 17. Στα τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά αποχές <clears throat> δεκτό. Τρίτο τμήμα υπέρ κατά αποχές δεκτό. Παράγος 19 σε έξι τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές δεκτό. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές δεκτό. Τρίτο τμήμα υπέρ κατά Φαντάζομαι ότι απορρίπτεται. Αρχίζουμε την ψηφοφορία ελέγχου για το τρίτο τμήμα. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίθηκε όμως. Τέταρτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Πέμπτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Με την προηγούμενη πλειοψηφία. Έκτο υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 22 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 25 μονομαστική κλίση αρχικό κείμενο έλεγχος 22 δεύτερο τμήμα βεβαίως άρχεται η ψηφοφορία ψηφίσατε όλοι πέρας εγκρίνεται 25 αρχικό κείμενο ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. 27 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 28 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 39 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 42 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. 39 έλεγχος ηλεκτρονικός άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίθηκε. 42 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 40 42-2 έλεγχος αρχή του ψηφοφορία ψηφίσατε όλοι πέρας απορρίπτεται 49 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 53. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 54. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 55. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές δεκτό. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 56. 55 δεύτερο τμήμα έλεγχος άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. 56 υπέρ. Κατά. Απόχες εγκρίνεται. 57 υπέρ. Κατά. Απόχες εγκρίνεται. 63 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 65 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 66 μονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία Abgestimmt. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. 67 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη D. Σε δύο τμήμα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτό. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτό. Αιτιολογική σκέψη I. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτό. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτό. Αιτιολογική σκέψη T. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αγαπητοί συνάδελφοι, πρωτού κάνουμε την τελική ψηφοφορία, θέλω να σας ζητήσω την επίοικιά σας, αν έκανα μερικά λάθη, αλλά προσπάθησα να έχω τη βοήθεια των ομάδων. Λοιπόν, είναι τελική ψηφοφορία επιτέλους. Ονομαστική ψηφοφορία και Αφήστε τις ε, κάρτες μέχρι να τελειώσει η ψηφοφορία παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Τα πρακτικά της συνεδρίασής μας θα εγκριθούν από το Κοινοβούλιο στην επόμενη συνεδρίωσή μας εάν δεν υπάρχουν καθόλου ε, αντιρρήσεις τα ψηφίσματα αυτά τα οποία έχουν εγκριθεί θα διαβιβαστούν στους αρμόδιους αποδέκτες. Δεν βλέπω καμία αντίρρηση. Διακόπτεται η συνεδρία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας εύχομαι καλή επιστροφή στις εστίες σας, καλή όρεξη.